Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Το und der Της ημερησίας διάταξης είναι η δήλωση για την συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμφουλίου. Το λόγο θα πρέπει να πάρει ο κύριος Φαν Ρομπόη, αλλά απουσιάζει. Άρα πρέπει να τον περιμένουμε.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 και εγώ μπορώ να σας διηγηθώ διάφορα για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, άμα θέλετε να ακούσετε δικά μου σχόλια, αλλά... Α, ωραία, ωραία, ωραία. Bonjour Monsieur le Président, bienvenue. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλώ ορίσατε. Είχαμε ξεκινήσει τη συνεδρίαση και έχετε το λόγο Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εξότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1η και 2η Μαρτίου ήταν